Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτα έκθεση Κόβατσικ. Η κυρία Πιετικάινεν. Η κυρία Πιετικάινεν. Η κυρία Πιέτη Κάινεν δεν είναι εδώ. Γιάρ, κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα εύκολα γιατί το θέμα είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τα αποθέματα μου. Αυτό το οποίο επίσης ήταν σημαντικό για εμένα είναι πως τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται μονίμως να τηρήσουν αυτές τις διατάξεις. Και αυτό το οποίο προξένησε έκπληξη ήταν και η συμπερίληψη της αλληλείας αναψυχής. Γιατί ακούγεται κάτι χαλαρό, έτσι αναψυχή, αλλά η αλληλεία αυτή έχει διαστάσεις επαγγελματικές πλέον. Και τέλος, Ευχαριστώ τα κράτη-μέλη τα οποία φροντίζουν για την σταθεροποίηση των αποθεμάτων μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ακολουθεί η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων μου από το Βορρά. Στην περιοχή της Βαλτικής υπήρξε υπερεκμετάλλευση των αλλιευτικών αποθεμάτων θεμάτων μπορεί αυτό να οδηγήσει σε εξαφάνιση των Σολομών και θα περιορίσει τη δραστηριότητα των αλλιέων. Γι' αυτό υποστηρίζω ένα πολιετές σχέδιο για την διαχείριση των αποθεμάτων Σολομού στη Βαλτική. Η Κομισιόν θα πρέπει να έχει αυστηρότερους ελέγχους στην αλλία αναψυχής ώστε να μπορέσει να ανακάψει το απόθεμα Σολομών στη Βαλτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακοβέη. Παρακαλώ, παρακαλώ όλους αυτούς που είναι ακόμα παρόν, κύριοι Μπροκ, Λίζε, Κασπάρη, Ρόουτσεκ, σας παρακαλώ. Είτε να ε, αποχωρήσετε ή τουλάχιστον να ακούτε, να είσαστε εδώ ήρεμοι και να ακούτε τις... Ε, επεξηγήσεις ψήφου. Κυρία Φερνίκη για την έκθεση Lightfried τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αφαίρεση των ε, πτερυγίων είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για ορισμένα είδη καρχαρίων. Έχει οικονομικές επιπτώσεις αλλά και από πλευράς ε, δεοντολογικής ε, δείχνει απόλυτη απουσία για τον σεβασμό της ζωής ε, των ζώων. Από μια πρακτική που ξεκίνησε το 2003 η Κομισιόν αποφάσισε να παρουσιάσει μια πρόταση η οποία στοχεύει στο να καταργήσει και την απαγόρευση εξαγωγή... αφαίρεσης των πτερυγίων στα αλληλευτικά σκάφη της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στους, ε, προσφέρουμε στους καρχαρίες την απαραίτητη προστασία, διότι αυτή η τεχνική η οποία εφαρμόζεται τώρα και στα ευρωπαϊκά ληφτικά σκάφη για την αφαίρεση των ε, πτερυγίων είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την ε, διαβίωση των ζώων και την δυνατότητα επιβίωσης τους. Κυρία Μακοβέη τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι επιτρέψει στην Κομισιόν να να εγκρίνει μη νομοθετικού χαρακτήρα πράξεις. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να τεθούν, να προσαρμοστούν αυτά τα, αυτοί οι κανονισμοί στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Η, η πρόοδος μας στα εμπορικά θέματα απαιτεί τη δυνατότητα της Κομισιόν να εγκρίνει μη νομοθετικές πράξεις. Αυτό θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και αυτό είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι όλα τα κατημέρια θα τηρήσουν αυτούς τους κανονισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέη, κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση διότι η κοινή εμπορική πολιτική επέτρεψε στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στους παραγωγούς να ε, έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Αυτή η πολιτική για να είναι αποτελεσματική η Κομισιόν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τροποποίησης κάποιων ουσιοδών κανόνων μέσω των πράξεων κατεξοδότηση. Στηρίζω τον εισηγητή, ο οποίος προτείνει πως ανα πάσα στιγμή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί σε θέματα που αφορούν ουσιώδη ε, σημεία της, ε, του, κανονισμού. Και η χρησιμοποίηση αυτών των πράξεων κατεξουδότηση θα πρέπει να γίνεται ε, με σωστό τρόπο και θα μπορείς να βοηθήσει στο να μην περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέη. Η αληθική πόρη είναι περιορισμένη πόρη, γι' αυτό τα μέτρα τεχνικής ε, διατήρησης είναι κέρια στοιχεία μιας προσέγγισης στη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων και πρέπει να έχουμε μια περιφερικοποιημένη αντιμετώπιση. Εγώ καταγράφω την πρόταση Κομισιόν, η οποία επεκτείνει τους κανόνες για τεχνικά μέτρα για μια περαιτέρω μεταβατική περίοδο που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να γίνουν οι επικαιροποιήσει. Υπάρχουν περιοχέ όπου απαγορεύεται η αλία σκόμβρου, βακαλάου και άλλων ηθίων. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει σαφήνεια σε σχέση με τις αλληλευτικές δραστηριότητες, ώστε οι ε, αλληλείς να βασίζονται σε μόνιμα και όχι προσωρινά μέτρα. Ζητώ από την Κομισιό να υποβάλει μια μόνιμη λύση για τα τεχνικά μέτρα το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες το βράδυ συζητήσαμε για τις συστάσεις αυτές που αφορούσαν τον αλληλευτικό τομέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήμασταν εδώ. Υπήρξε λοιπόν αυτή τη ευρύτατη συζήτηση και όλα αυτά με ενθαρρύνουν γιατί δείχνουν ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι σοβαρές, πρακτικού χαρακτήρα και ιδίως θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τον Πάτ Κόμπ Γκάλαχερ, τον Ιρλανδό συναδελφό μου, για την δική του εργασία. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να δεχτούμε στην τελευταία ψηφοφορία ορισμένες συστάσεις, γιατί δεν υπήρξε πραγματική συνεργασία από την πλευρά του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Και είχε μεγάλο δίκιο ο κύριος Γκάλαχερ όταν ζήτησε την αναβολή της τελικής ψηφοφορίας γιατί μόνο με κάποια συνεργασία του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Πατράου, έκθεση Πατράου Νέβες, η κυρία Πιετικά είναι, αλλά δεν εδώ η κυρία Πιετικά Πιετικά, η κυρία Μακλάρκιν έχει το λόγο. Η αποκοπή των πτεργείων των ε, καρχαριδών είναι μια πρακτική που δεν μπορώ να υποστηρίξω ούτε και η πολιτική μου ομάδα. Οποιαδήποτε παρέκκληση από την νομοθεσία που επιτρέπει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να σταματήσει παρά αυτά. Είναι μια βαρβαρική πρακτική που οδηγήσει σε θάνατο, ε, από πνιγμό ή από ασυτεία των καρχαραϊδών. Είναι μια ντροπή να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ε, πλάσματα με αυτόν τον τρόπο. Παραβιάζει κάθε μορφή ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ζώων και είναι έσχος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει άλλες χώρες στον κόσμο ε, αλλά όχι τον εαυτό της για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Δεν πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να αφήσουν να, γίνει, να γίνεται εκφόρτωση των ε, ηχθείων αυτών χωρίς τα πτερυγιά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μακλάρκιν. Η κυρία Γετζέσκα έχει τώρα το λόγο. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για την βαρβαρική αυτή πρακτική της αποκοπής των πτεργίων. Αυτή η πρακτική είναι μια βάρβαρη πρακτική, είναι σπατάλη και ε, στρέφεται κατά της διατήρησης αγρίων ειδών, ειδών. Γι' αυτό εγώ υποστήριξα αυτήν την ε, έκθεση και ζητώ την απαγόρευση αυτής της πρακτικής χωρίς την παραμικρή εξαίρεση. Θα πρέπει να κλείσει τα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν οι Κομισιόν για την αποκοπή των πτερυγίων και θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Είναι μια πρακτική η οποία εφαρμόζεται πολλές φορές στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Αυστραλία. Αλλά τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να στραφούν εναντίον της και να αποφύγουν οποιαδήποτε παρέκκληση. Ευχαριστώ. Κυρία Γιατζέσκα. Η κυρία Τσανίκη νομίζω ότι έχει φύγει. Ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά μπορέσα εγώ να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση γιατί εδώ και 10 χρόνια διεκδικεί η δική μου πολιτική ομάδα αυτή την προστασία και στη γερμανική Bundestag έχουμε επιτύχει να έχουμε μια απαγόρευση αυτής της βαρβαρικής πρακτικής και τώρα έχουμε μια ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποκλεί κάθε παρέκκληση ακόμα και αν είναι καλής πρόθεσης. Μια τέτοια πρακτική είναι βαρβαρική, δεν είναι ηθική και θα πρέπει να καταργηθεί στο όνομα της προστασίας των ε, ζωικών ειδών. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ούτε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο να γίνεται παραδεκτή αυτή η πρακτική. Ξέρουμε ότι είναι απαράγραπτη η ανάγκη προστασίας των θαλασσίων ειδών και νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία ψήφιση αυτής της ε, έκθεσης. Σας ευχαριστώ, ε, κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις καρχαρίες αλλά οι καρχαρίες βρίσκονται στον κόσμο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς αιώνες. Και σήμερα εμείς μιλήσαμε και για την υποστήριξη των καρχαραϊδών όταν απαγορεύσαμε την πρακτική του λεγόμενου φίνινγκ, την αποκοπή των πτερίγιων. Μπορεί αυτό να θεωρείται λιχουδιά για πάρα πολλούς, το πτερίγιο του καρχαρίου. Αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκόπτονται τα πτερήγια και να απορρίπτονται οι καρχαρίε στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι μοναχαβαρβαρικό, είναι μια πραγματική σπατάλη και είναι αρνητικά πολύ τα αποτελέσματα αυτά για τους καρχαρίες που μετά χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται λοιπόν αυτή η πρακτική. Είναι θετικό ότι σήμερα καταφέραμε με μεγάλη πλειοψηφία να τονίσουμε ότι αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι απαγορεύσεις οι, οι μάλλον θα πρέπει να απογορευτούν και πρέπει οι καρχαρίε να εκφορτώνονται ολόκληρε στι ακτέ. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μακοβέη και πάλι. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω το νομοθετικό ψήφισμα για την πρόταση εντροπής του κανονισμού 1113 ε, ε, ε, του Συμβουλίου και ε, Επιθυμούμε να απαγορευτεί πλήρως, ε, δίχως ε, παρεκκλήσεις, ε, η αφαίρεση των πτερυγίων στα σκάφη τα Παρόμοια πρακτική, δηλαδή η αποκοπή των πτερυγίων και η απόρριψη του σφάγιου στην θάλασσα είναι μια φοβερή πρακτική, πρέπει να απαγορευτεί απανταχού. Tannock. Κύριε Πρόεδρε, η αφαίρεση των πτερυγίων από τους Καρχαρίας είναι μια βάρβαρη πρακτική. Συμφωνώ την εκστρατεία που έχει αναλάβει η οργάνωση για την προστασία των ζώων σχετικά με την ε, αποκοπή των πτερυγίων και τη χρήση τους για την Παρασκευή Σούπας. Έφτασε Χρόνο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προωθήσει αυτή την απαγόρευση και να ακολουθηθεί από άλλους ε, χώρες. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της υπεραλίευσης ορισμένων ε, ειδών καρχαρία, κάτι το οποίο απειλεί με εξαφάνιση τα είδη αυτά. Πρόκειται για, ένα, για είδη τα οποία ζουν στις θάλασσές μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο συνάδελφος Μπέρφη για να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την περιορισμό των ε, κενών που υπάρχουν σε αυτόν τον κανονισμό προκειμένου να απαγορευτεί η αφαίρεση των ε, πτερυγίων, των καρχαριών ε, στα αλληλευτικά σκάφη. Αυτό δεν έχει καμία, σχέση, καμία θέση συγγνώμη, στην σημερινή πρακτική αλίας. Καταδικάζουμε τους καρχαρίες σε έναν επίπονο θάνατο. Είναι μια πρακτική η οποία εφαρμόζουν διάφορες πολυεθνικές εταιρείε. Δέκα εκατομμύρια καρχαρίες υπολογίζεται ότι φωνεύονται ετησίως και αυτό όπως καταλαβαίνετε οδηγεί σε δημιουργία μιας αστάθειας στον ζωικό θαλάσσιο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μέρφυ. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για τα θέματα απαγωγής ε, παιδιών. Η κυρία Μουσκαρδίνη έχει το λόγο. Πρόεδρο, είμαστε υπέρ του ψηφίσματος που υπερψηφίστηκε σήμερα για το θέμα της απαγωγής ε, των παιδιών. Το πρόβλημα όμως ε, συνεχίζει να υφίσταται στα κράτη-μέλη. Κανείς, ε, όχι όλοι, δεχτήκαν την εφαρμογή του και συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες το και Jugendamt στην Γερμανία όπου τα δικαιώματα των παιδιών τίθενται σε δεύτερο επίπεδο Ελπίζουμε με το ψήφισμα αυτό να ε, οδηγήσει σε μια βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει αυτό να αποτελεί προτεραιότητα των κρατών μελών και να ε, οθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη συνθήκη της, τη σύμβαση της Χάγης, να βρουν τη σωστή ε, ισορροπία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό θεσμός για το οικογενειακό δίκαιο. Ευχαριστώ κύριε Μουσκαρδίνη. Κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ. Η διεθνή απαγωγή παιδιών είναι μια τακτική η οποία θα μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Η σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα περί απαγωγής παιδιών επιθυμεί να ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Το Συμβούλιο αμφισβητεί την, βάση, την νομική βάση προκειμένου να συμπεριληφθούν οκτώ νέα μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουμε κάτι προσπάθεια. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ε, δεχθεί περαιτέρω καθυστερήσει. Ε, ζητούμε ε, από την Επιτροπή να διευκρινίσει το συντομό των δυνατών την, ευρωπαϊκή, την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα θέματα που αφορούν την διεθνή απαγωγή παιδιών. Κάθε λεπτό που περνάει, κάθε ώρα που περνάει είναι εις βάρος ε, της ε, κατάστασης των παιδιών. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Έχουμε κλείσει με αυτό το θέμα. Ερχόμαστε στις ε, ταξίες ψήφου για τη διάσκεψη της Ντόχα. Η κυρία είναι δεν είναι παρούσα, η κυρία Ζαμπόσκα έχει το λόγο. Ναι, ναι, έχετε το λόγο. Για την Δόχα. Doha, Doha. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το ψήφισμα. Δεν το υποστηρίξα γιατί έλαβαν υπόψη την συμμετοχή της Σλοβακίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών. Οι χώρες μας έχουν τηρήσει τα υπεσχημένα φάση του πρωτοκόλλου του Κιωτό και έχουν βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει στο προσκήνιο του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Είναι απαράδεκτο η συνεισφορά των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα πρέπει η τα πιστοποιητικά εκπομπών να μεταφέρονται από τις χώρες αυτές αλλού και όλες αυτές οι απαγορεύσεις θα εμποδίσουν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Σλοβακίας να συμμετάσχουν στην πράσινη οικονομία. Σας ευχαριστώ κυρία Σαμπόρσκα. Η κυρία Μπασέσκο ακολουθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να υπερσφίσω το ψήσμα διότι η Ρουμανία δεν έχει φτάσει ακόμα στην απαραίτητη ποσόστοση και έχει ακόμα πολλά διαθέσιμα πιστοποιητικά. Ε, επειδή τα πιστοποιητικά αυτά δεν μπόρεσαν να τύχουν εμπορίες, κινδυνεύουμε να απολέσουμε πολλά ε, σημαντικά ποσά. Για το πιστεύω ότι τα κράτη που έχουν διαθέσιμες ποσοστώσεις να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασία του περιβάλλοντο. Με τι δεσμεύσει που έχει λάβει η Ρουμανία στο πλαίσιο τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, ε, δείξαμε την δέσμευσή μα ε, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά απαγορεύοντα τη μεταφορά ποσοστώσεων για μετά το 2012, το, η χώρα μου υφίσταται ε, διακριτική μεταχείριση σε σχέση με άλλα κράτη που βρίσκονται στην αυτή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τις τηλεπικοινωνίες και εδώ πέρα θέλει η κυρία Μπασέσκου να κάνει ξανά μια επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι υποστηρίζω την αναθεώρηση του Διεθνού Κανονισμού για τι τηλεπικοινωνίε που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τη διασκέψεω. Στόχο είναι να διευκολύνει την διεθνή διασύνδεση των υπηρεσιών και των ε, πληροφοριών ε, αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Ε, χρειάζεται λοιπόν να καταστούν οι υπηρεσίε αυτέ αποτελεσματικέ. Πρέπει να διασφαλίσουμε την κυκλοφορία αυτών των πληροφοριών Θεωρώ ότι το κείμενο του κανονισμού χρειάζεται να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να αντανακλάμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αλλαγές στην τεχνολογικό τομέα. Η διάσκεψη αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη και μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη για να πετύχουν νέα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ε, και να ανταποκριθούμε με καλύτερε προκλήσει του περιβάλλοντος που εξελίσσεται άρδιν. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Περνάμε στην έκθεση ΚΟΠΑ. Πρώτη επεξήγηση ψήφου η κυρία Νικολάη. Ε, Υπερψήφισα αυτή την έκθεση της κυρίας Κοπά δεδομένου ότι το κείμενο θέλει να δημιουργήσει μια... το κείμενο από το κείμενο διαγράφηκε η δημιουργία νέας ε, κατηγορίας ε, μελών. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την ε, προσπάθεια διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει, αποτελεί μια θετική νότα, μια αισιόδοξη νότα, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε τις επιτυχίες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια της Κοπεχάγης ε, παραμένουν σε ισχύ. Εξετίμησε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η κυρία εισηγήτρια αντιμετώπισε το ζήτημα των ικανοτήτων των νέων υποψηφίων χωρών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για να μην μπλοκαριστούν οι ιστορικοί μηχανισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στάτλερ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την έκθεση ΚΟΠΑ γιατί πρώτα απ' όλα ζητάει την ανεφόρον στήριξη του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης και δεν αναφέρει ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Αναφέρει μάλιστα και θετικές εξελίξεις στην Τουρκία. Μα δεν αναφέρει πως μέχρι σήμερα διώκονται εθνοτικές μειονότητες, θρησκευτικές μειονότητες και ειδικά οι χριστιανοί και για πολλωστή φορά ο Τούρκος Πρωθυπουργό, ο Ερντογάν, ε, μίλησε για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Ποιες είναι οι θετικές εξελίξεις, δηλαδή δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Ψήφισα από βαθύτατη πεποίθησή μου κατά αυτής της έκθεσης, η Τουρκία δεν είναι όριμη για την Ευρώπη και δεν θα ενταχθεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι την ε, τωρινή αυτή ε, διεύρυνση η ένταξη στην Ευρώπη σήμαινε βελτίωση της ασφάλειας των χωρών και της οικονομικής τους κατάστασης ε, ειδικά, κατάστασης ειδικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως αυτός των Βαλκανίων. Ελπίζω λοιπόν σύντομα και η Κροατία να ενταχθεί και να ακολουθήσουν και οι γειτονές της. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει, όπως είπαμε, και η διεύρυνση προς Ανατολάς. Για την Πολωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ουκρανία, ο μεγάλος μας γείτονας. Πρέπει επίσης να δώσουμε κίνητρα στην νέα κυβέρνηση της Γεωργίας για να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πορεία. Η στήριξη της διεύρυνσης είναι κάτι το επιθυμητό και ε, συμφωνεί με αυτά τα οποία θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Μπιέλεν. Η κυρία Μακοβέη. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πολιτικέ διεύρυνση και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ραμμένα και κομμένα στι ικανότητε και δυνατότητε των κρατομελών και των πολιτών. Για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο ικανοποιητικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταρρύθμιση στον δικαστικό τομέα και την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Ε, χαιρετίζω την πρόληψη της Κομισιόν για να ανοίξει τα κεφάλαια 23 και 24 στα διαδικασία ε, προσχώρησης. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ότι η πλήρωση αυτών των ε, προϋποθέσεων είναι απαραίτητο. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να, τα κριτήρια να είναι διάφανη. Το ζήτημα της, ε, των, των διαπραγματεύσεων με την Μακεδονία θα πρέπει να μας ε, οδηγήσει στο να προτείνουμε την έναξη διαπραγματεύσεων τώρα. Ευχαριστώ. κυρία Σμόλκοβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. We have to, πρέπει να ε, τονίσουμε την σημασία των κριτηρίων της για τα κράτη που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κάθε κρίση οδηγεί και σε νέες αξίες σε νέα στοιχεία αλληλεγγύης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές προκλήσεις που είναι πολύ σημαντικές. Πολλοί από εμά δεν θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη διαδικασία διεύνησης που έχει συμβάλει στην ειρήνη, σταθερότητα της, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Υπήρου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου που είναι η βάση της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε, χάρη στη διεύνηση, να ξεπεράσουμε τους διχασμούς του παρελθόντος και να αναλάβει και η Ευρώπη ένα σημαντικότερο ρόλο στο διεθνές στερέωμα και θεωρούμε λοιπόν ότι η διαδικασία διεύνηση θα βασίζεται σε μια διάφανη και ε, σαφή σειρά κριτηρίων που δεν θα επιδέχονται ερμηνείες και θα είναι καταμετρήσιμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σμόλκοβα. Τελευταίος ομιλητής για την έκθεση αυτή ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κυρίας Κοπά δεν είναι κακή, αλλά έχει βασικά προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Μακεδονία χρειάζεται τη συζήτηση υψηλού επίπεδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να ε, συνοδεύεται από την άρση του ελληνικού βέτο εναντί της ε, Μακεδονίας. Για το κοσφοπέδιο παραμένουν οι υποσημειώσεις οι οποίες πολλές φορές συνοδεύουν τη χώρα αυτή, αλλά είναι μια ανεξάρτητη χώρα η οποία είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει οι πέντε χώρες οι οποίες θα την υποσημειώσει και οι οποίες αρνούνται να αναγνωρίσουν το κοσφοπέδιο να αλλάξουν γνώμη και να κατανοήσουν ότι αυτή η χώρα βρίσκεται πια στα πλαίσια μια συμφωνία εμπορική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο. και εγώ θέλω να καταδικάσω την εφημιστική διατύπωση που χρησιμοποιείται για την Τουρκία. Ήταν ένα λάθος να θεωρηθεί η Τουρκία ως υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι Ευρωπαϊκή χώρα και δεν εκπληρεί τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Αυτά για την έκθεση ΚΟΠΑ. Ακολουθεί η ακολουθούν οι επεξηγήσεις ψήφου για την κατάσταση στην Γάζα. η κυρία Κοστέλλο. Σας ευχαριστώ κύριε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την κατάψη του πυρός που ανακοινώθηκε χθε στην Γάζα και καλό για μια πλήρη εφαρμογή του και από τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ε, φεύγουν βλήματα από πλευρά της Γάζης ε, αλλά και οι Ισραηλοί θα πρέπει να πάψουν τους βαρδιμούς της ε, Γάζας και τις δολοφονίες αξιωματούχων. Διαφορετικά σε μερικούς μήνες θα ξαναμαστε πάλι εδώ και θα συζητάμε το ίδιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν προσυπέραψα και υπερψήφισα το ψήφισμα όπου καλούμε να πάψει ο αποκλεισμό της Γάζας μεταξύ άλλων να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των Παλαιστινιακού λαού να ζήσουν ειρηνικά εντός των σύνορων. Ικανοποιήθηκα από το ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη να καταστεί η ε, Παλαιστινιακή Αρχή ε, παρατηρητής στον ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κοστέλο. Ο Μπίλ αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, βεβαίως σύγκρουση ποτέ δεν είναι επιθυμητή. Όταν μιλάμε για την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολή. εμείς έχουμε υποστηρίξει τη συνύπαρξη των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, ως ε, δύο ανεξάρτητων κρατών. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες για την ασφάλεια σε αυτή την περιοχή, όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή μας αναγκάζει να απευθύνουμε ξανά έκκληση για να σταματήσει η βία και πρέπει να καταδικάσουμε και τις επιθέσεις με ρουκέτες της ε, Χαμάς και το λαθρεμπόριο όπλων προς τους Παλαιστινίους και η κυβέρνηση στο Τελαβίβ αναγκάστηκε να υπερασπιστεί κατόπιν την χώρα της ε, απέναντι στην επιθετικότητα της ε, Παλαιστίνης. Εγώ στηρίζω το ψήφισμα και είμαι υπέρ της λύσης δύο ανεξαρτήτων δημοκρατικών κρατών. Όμως ε, καταδικάζω τις ε, πράξεις των ε, ακραίων Παλαιστινίων και την άρση του αποκλεισμού της Γάζας. Ευχαριστώ. Κύριε Στάντλερ, κύριε Πρόεδρε, εγώ ψήφισα αυτό το ψήφισμα και δεν πάει αρκετά μακριά κατά την απόψή μου. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα πως τα 600 εκατομμύρια ευρώ που στέλνει στην περιοχή κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνδεθούν με όρους και για τις δύο πλευρές. Αυτά τα οποία είπαμε βεβαίω ισχύουν και για τις δύο πλευράς ε, εξίσου. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο Ισραήλ πως ε, πρέπει να δει το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει κανείς για πάντα τους ανθρώπους πίσω από ένα σειρματόπλεγμα και ένα τείχος. Δεν είναι ε, πράγματα αυτά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συνομιλήσουν με την Χαμάς. Οι Αυστριακοί έχουν ε, μεγάλη παράδοση ως ε, διαμεσολαβητές. Μας είχαν ασχίσει κριτική όταν μιλήσαμε με τον Ραφάτ, αλλά αποδειχθήκαμε σωστή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και σήμερα. Ευχαριστώ η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι Ικανοποιημένη για το ότι μπορέσαμε να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα για την Γάζα όπως ε, πολλοί συνάδελφοι έτσι και εγώ είμαι ικανοποιημένη για την κατάβαση του πυρός. Όμως δεν μπορούσα να στηρίξω το άρθρο 5 του προτινόμενου ψηφίσματος, το οποίο ξεπερνάει την φύση του ψηφίσματος. Αν είναι να μιλάμε για συμβαστική λύση αποδεκτή και στις δύο πλευρές, δεν πρέπει μονομερώς να στηρίζουμε ε, αυτά τα οποία ισχυρίζεται η μία πλευρά. Δεν είναι ισορροπημένη προσέγγιση αυτή, δεν θα βρούμε έτσι ειρηνική λύση. Η κρατική κυριαρχία της επικράτειας των Παλαιστινίων ε, ε, πρέπει να είναι ανταμοιβή και όχι προϋπόθεση για τις προσπάθειές τους να ζήσουν εν ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέρφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για κατά τη διάρκεια 8 ημερών ο λαός της Γάζα της Γάζας είχε να αντιμετωπίσει μια τρομερή επίθεση από το Ισραήλ. Χάσαν τη ζωή τους τουλάχιστον 150 Παλαιστίνοι, οι περισσότεροι άμαχοι και πολλοί από αυτούς παιδιά. Από πολλούς ε, βραβευμένους με το βραβείο Νόμπελ, από τον Ομπάμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε τη συνηθισμένη υποστήριξη για την αφήγηση του Ισραήλ, ότι δηλαδή έχει το δικαίωμα να προστατεύσει τον πληθυσμό τους, όπως είπαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως η επίθεση με την ασφάλεια των Ισραηλινών. Είχε να κάνει πολύ με το κατεστημένο, το δεξί κατεστημένο, το δεξιά πτέρυγα του κατεστημένου στο Ισραήλ που θέλει να εμποδίσει οποιαδήποτε βοήθεια να υπάρξει αναγνώριση από τον ΟΗΕ για την Παλαιστίνη. Εγώ χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο λαός της Γάζας να είναι ήσυχος, ότι θα ξαναβομβαρδιστεί. Μια πραγματική όμως η ειρήνη θα απαιτήσει το τέλος της καταστολής του λαού της Παλαιστίνης και μια αλλαγή του καθεστώτος στην περιοχή προς το συμφέρον της εργατικής τάξης. Το Ισραήλ μπορεί να το κάνει αυτό μόνο άμα δεχτεί την πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριε Μέρφυ. Η κυρία Μόρκου Νάιτε Νικουλένιε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να υποστηρίξω τους συναδέλφους οι οποίοι χαιρέτησαν την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι μια συμφωνία που θα διαρκέσει και θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις ειρήνης για το, την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών στην περιοχή. Το ψήφισμα είναι εξισορροπημένο. Αναφέρει την ε, λύπη μας για τον θάνατο των αμάχων, καταδικάζει τις ε, επιθέσεις και κατά των αμάχων στο Ισραήλ, αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ, αλλά οποιασδήποτε προσπάθειες που γίνονται για να στοχευτεί ο άμαχος πληθυσμός δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αναφέρεται επίσης το ψήφισμα για την αίτηση του, των Παλαιστινίων να γίνουν παρατηρητές στον ΟΗΕ. Υποστηρίζουμε την ε, δημιουργεί ενός κράτους για την Παλαιστίνη, αλλά πρώτα θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Παλαιστινίου και Ισραήλ για να εισέλθει στον ΟΗΕ η Παλαιστινιακή Αρχή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η λίστα βρεθεί επί τη βάση της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ευχαριστούμε κυρία Μορκουνάιτε. Ακολουθεί ο κύριος Πόσελτ. Για την ε, κατάπαυση του πυρός στην ε, Γάζα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι και κημητήριο ανακοχών η περιοχή της Παλαιστίνης. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μία μόνιμη λύση για την περιοχή αυτή και αυτό δεν μπορεί να βασιστεί σε τίποτα άλλο παρά μόνο πάνω στο δικαίωμα ε, επιβίωσης του Ισραήλ και των, μέσα σε ασφαλή σύνορα από τη μια μεριά και το δικαίωμα από την άλλη πλευρά να έχουν οι Παλαιστίνοι το δικό τους κράτος μέσα σε μια λύση στο δικαιωμα επιβιωσης του ισραηλ και τον μεσα σε ασφαλη συνορα απο τη μια μερια και το δικαιωμα κρατών. Παρά το γεγονός ότι αυτό αναφέρεται σωστά στο σημείο 30 του ψηφίσματος, ε, εγώ δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω το σημείο 5 ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί εν καιρό η Παλαιστίνη στις δομές του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάτι τέτοιο και μια τέτοια δήλωση θα ήταν λαθασμένο μήνυμα όταν η περιοχή αυτή που ελέγχεται από την Χαμάς έχει στείλει εκατοντάδες πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Πρώτα μια ειρηνική λύση και μετά η ενσωμάτωση της δομές του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί για την ε, έκθεση αυτή κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Απήχα τις ψηφοφορίες διότι ακόμα και αν είμαι υπέρ της ε, διαδικασία ειρήνευση, δεν θεωρώ ότι η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί ενώ η Χαμάς διαλέγει την βία και όχι τον δρόμο της διαπραγματεύση Τώρα, σε ό,τι φορά το ζήτημα του ε, καθεστώτος παρατηρητή στον ΟΗΕ, νομίζω ότι αυτό θα επιδεινώσει περαιτέρω την στάση της Χαμάς στο Ισραήλ. Φυσικά έχει το δικαίωμα να προστατεύει το έδαφο την επικράτειά του, αλλά δεν ε, ε, και να μην επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να δολοφονούν αθώους. Η βόμβα η οποία εξεράγει στον ε, Τελαβή προχθές δείχνει τις προθέσεις της Χαμάς. Η Χαμάς ε, χρειάζεται να σταματήσει αυτές τις στρατιωτικές επιθέσεις και να σεβαστεί την συμφωνία περί καταπάψης του πυρός που ανακοινώθηκε χθες. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Έχουμε κλείσει τις ε, επεξηγήσεις για την κατάσταση στη Γάζα. Περνάμε στην ε, επεξηγήση για την έκθεση Νταουζάν με τον κύριο Στάντλερ. Έχω καταψηφίσει αυτό, το, αυτή την έκθεση, κύριε Πρόεδρε, γιατί εγώ δεν μπορώ σαν εκπρόσωπο Αυστρία να δεχτώ αυτά τα οποία αναφέρονται. Όλα αυτά οδηγούν σε μια περαιτέρω στρατικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν αναφέρεται τίποτα για μια διαδικασία πυρηνικού ε- αφοπλισμού. Θέλουμε την στρατιωτική συνεργασία μονάχα με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ουσιαστικά η διάκριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Για μένα, σαν εκπρόσωπο μιας ουδέτερης χώρας, αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι αυτή δεν μπορεί να υποστηριχθεί η έκθεση αυτή από εκπροσώπους της δικής μου χώρας και από άλλους βουλευτές αυτή της ε, Ολομέλης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την έκθεση Ντονζόν γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις στρατηγικές τους δυνατότητες και τις ε, δυνατότητές τους μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ε, ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της κρίσης και να αναπτυχθεί στην πλήρη ικανότητά, τους, ικανότητά της, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς που εισάγονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης το σημαντικό ρόλο των στρατιωτικο-πολιτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως παράδειγμα, στο πλαίσιο αυτό, θέλω να αναφέρω τη μεγάλη μας αποστολή στο Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κούκαν. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεξάγει 19 ε, πολιτικές αποστολές και 20 στρατιωτικές. Έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε στη σταθερότητα στα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Έχουμε συνεισφέρει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Σήμερα τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά το κράτο δικαίου, προστασία μειονοτήτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορέσει να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις και τις γεωπολιτικές αλλαγές στη διεθνή σκηνή. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε ξανά την στρατηγική μας, να είμαστε πιο αυτόνομοι και να δείξουμε περισσότερη ενότητα. Μεγαλύτερη εξαρτησία δεν σημαίνει πως οι υφιστάμενες συμμαχίες θα παραμεληθούν αντιθέτως, θα ενισχυθούν οι ισχυρές διατλαντικές σχέσεις. Έχει φτάσει η ώρα για μια φιλόδοξη και πάμε τα ανάλογα μέσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση γιατί θεωρώ πως ε, η στρατηγική ασφάλειας του παρελθόντος δεν επαρκεί δεδομένων των νέων προκλήσεων ασφαλείας παρά το ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από κάποια κράτη-μέλη που επηρεάζονται από την κρίση και έχουν χαμηλού προπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο για να διασφαλίσει την ασφάλεια των καρτομελών και των πολιτών του. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να επαναφέρει την στρατηγική της ανεξαρτησία μέσω μιας ισχυρής και ανεξάρτητης ε, ΚΕΠΑ για να μπορεί να δράσει ανεξάρτητα. Έχουν επηρεαστεί οι αμυντικές μας δυνατότητες από την οικονομική κρίση, αλλά η πολιτική της Ένωσης δεν πρέπει να αφαιθεί σε άλλους. Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Κομισιόν και Συμβούλιο πρέπει να ορίσουν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης και βεβαίως αυτό όχι μόνο για να διαφυλεχθούν οι ε, κοινότητε αυτέ τη ασφαλεία, αλλά για να μπορέσουμε και εμεί να αντιδράσουμε στι νέε αυτέ προκλήσεις. Σας ευχαριστώ, κυρία Σμόλκοβα, κύριο Στάνοκ, κύριε Πρόεδρε. Οι συντηρητικοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πολλές επιφυλάξεις για την ΚΕΠΑ, καθώς θα έχουμε επικάλυψη με το ΝΑΤΟ, το οποίο πρέπει να παραμείνει ο πυλώνα της Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ σημαίνει και ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και έχουμε σοβαρές ανησυχίες αποσύνδε, αποσύνδεσης από τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Θεωρώ όμως πως είναι στο συμφέρον της Βρετανίας να εμπλακεί ρεαλιστικά στις επιχειρήσεις όταν μπορεί να συνεισφέρει. Είμαι εισηγητή για το κέρα Αφρική και πρέπει να παραδεχτώ πω η αποστολή Αταλάντα αλλά και η εκπαιδευτική αποστολή στην Ουγγάντα είναι χρήσιμε. και θα παρακολουθήσω ε, την αποστολή στο Μαλί με ενδιαφέρον μαζί με την ΕΚΟΒΑΣ για να ειρνεύσουμε την περιοχή εκεί, καθώς επίσης και την αποστολή EULEX στο Κοσφοπέδιο, η οποία έχει αποδειχθεί ε, χρήσιμη. Παραμένω, όπως είπα, επιφυλακτικό, αλλά παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συμπληρώσαμε 90 ε, χρόνια από όταν ο Χόβε Καλέργης ε, έκανε την πρότασή του για μια πανευρώπη. Και βεβαίως μιλούσε για κάποιες ε, Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης και αυτός ο οποίος ήταν ειρηνιστής μιλούσε, εννοούσε μια κοινή αμυντική πολιτική και δυνατότητα επίλυσης διαφορών. Και είναι νομίζω στο πλαίσιο αυτής της παράδοσης που θα πρέπει η Ευρώπη να επικεντρωθεί στις βασικές της αρμοδιότητες και αν μου επιτρέπετε να αναφέρω δύο άλλους μεγάλους Ευρωπαίους, τον Ότο Φον ο οποίος φέτος θα συμπλήρουν τα 100 του χρόνια, και τον Φραντς Γιώζεφ Στράους, είπε πως το ΝΑΤΟ έχει μέλλον εάν στηριχθεί σε δύο ισοδύναμους εταίρους, τις ΗΠΑ Αμερικής και τις ΗΠΑ. της Ευρώπης. Αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό κάνει η έκθεση Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Ακολουθεί ο κ. Τσαρνέσκη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι επιφυλακτικός απέναντι στις, ε, σε αυτά τα οποία προσπαθούμε να ε, έχουμε ως βάση της ε, κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής Νομίζω ότι είναι αυτά που μακρύνονται από την πραγματικότητα. Πρόσφατα ε, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση. Οποιοδήποτε βασικό ζήτημα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική προκαλούσε διαφωνίες μεταξύ των μεγάλων κρατών μελών της Ένωσης. Και, και τώρα παρόμοια είναι η κατάσταση, γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, γιατί η δική μου εντύπωση είναι πως δεν χρειαζόμαστε μεγάλα λόγια και μοδάτα λόγια για την ε, διεθνή συνεργασία. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε την κοινή μας αμυντική πολιτική, βεβαίως. Σας ευχαριστώ κύριε Τσαρνέσκι. Αυτά για την έκθεση Ντόνζο. Ερχόμαστε στην έκθεση Πάσκου με την κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Επιθυμώ να σχολιάσω την έκθεση την οποία στήριξα, υπερψήφισα. Είναι μια έκθεση πολύ σημαντική στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας ε, και ασφάλειας. Η αλληλεγγύη και η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας ε, αναλύονται εδώ και ύπαρξη μιας ε, κοινή πολιτική υφίσταται, αλλά δεν υπάρχουν τα εργαλεία προκειμένου να ε, εφαρμόζονται στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι φορά τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα, η συνδρομή που προλείπεται από το άρθρο 30 τη ε, συνθήκη, η έκθεση προτείνει ένα στρατηγείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μόνιμο στρατηγείο, το οποίο θα δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει ενωμένη ε, την ρήτρα αυτή. Σε ό,τι φορά τώρα τη ρήτρα αλληλεγγύη. διακόπτη ο πρόεδρος τα μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Ο κύριο ε, Στάντλερ, κύριε πρόεδρε. Και εγώ καταψήφισα αυτή την έκθεση, όπω και την ε, εναντίον των εκθέσεων Κέλαμ και Τάρεντ για τους ίδιους λόγους, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο εκφράζονται και στην έκθεση Ντάμσον Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι η έκθεση αυτή είναι ασαφής σε δύο πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Τι θα πει η υποχρέωση να υπάρξει αρρωγή με κάθε μέσο. Αυτό ξεπερνά ακόμα και αυτά που λέει το ΝΑΤΟ. Είναι ιδιαίτερα ασαφής αυτή. Τι είναι ανθρωπογενής κρίση. Οποιαδήποτε κρίση μπορεί να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης. Αυτό για μια ουδέτερη χώρα είναι απόλυτα απαράδεκτο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ασάφεια σε αυτή την έκθεση, ιδίω για τα θέματα αυτά των καταστροφών που θα πρέπει να οδηγήσουν σε αρρωγή. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ εγώ να δώσω την έγκρισή μου σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Στάτλερ. Η κυρία Μακοέι. οποιοδήποτε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή ή να είναι θύμα μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε μεγάλη ταχύτητα σε τέτοιες κρίσεις και να υποστηρίξουμε τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξουν μια πολιτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων απειλών ασφάλειας. Καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να ημωγούμε εκ των υστέρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να, εξασφαλίσουμε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει φυσικά να βρούμε και τη σωστή ισορροπία που θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την λογοδοσία για τη λήψη αποφάσεων. Είναι κέρια η λογοδοσία. Σας ευχαριστώ κύριε Μαχοβέ, ακολουθεί κύριε Μπεζέσκου. Ευχαριστώ, υπερψήφισα την έκθεση διότι θεωρώ ότι για να προσδιορίσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα έχουμε ανάγκη από την ενίσχυση της κοινή πολιτικής άμυνας. Το τομέα της κοινή άμυνας η αλληλεγγύη ανάμεσα στα κρατημέλη είναι πολύ σημαντική. Αλλά αυτή η αλληλεγγύη θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλους μηχανισμούς χρηματοδότηση. Η ρήτρα αμοιβαίας ε, άμυνας ε, συνδρομή είναι ένα μέσο αποτελεσματικό εάν κάποιο μέλος ε, ε, γίνει αντικείμενο επίθεση. Δεν έχουμε προ το παρόν μια τακτική για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια ρήτρα. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί λοιπόν με τρόπο αποτελεσματικό η Κομισιόν θα πρέπει να οργανωθεί σε επίπεδο τόσο τεχνικό όσο και πολιτικό. Ακόμα και αν υπάρχει κίνδυνο ε, ένα κράτο μέλο να υποστεί επίθεση πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στι νέε απειλέ όπω η τρομοκρατία και οι επιθέσει στον κυβερνοχώρο. Αυτέ οι κατάσταση, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριοποίησης της ε, ρήτρα ε, αμοιβαία Άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Αυτά για την έκθεση Πάσκου. Για την έκθεση Κέλαμ. Η κυρία Αντεστότερ δεν είναι παρούσα. Η κυρία Νικολάη έχει το λόγο. Υπερψήφισα την ε, έκθεση την οποία θεωρώ ότι είναι η πρώτη και η πιο σαφής έκθεση που ασχολείται με την ασφάλεια των, του κυβερνοχώρου. Διότι οι υπόλοιπε παρεμβάσει που αφορούσαν ε, την προστασία του κυβερνοχώρου δεν ε, είναι εισάξιες και αντάξιες ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό αυτό των επιθέσεων ε, στον χώρο. Μόνο 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια εθνική στρατηγική ε, αντίδραση σε αυτές τις ε, επιθέσεις στον χώρο που αποκτούν όλο και περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Γνωρίζαμε καταστάσεις σε κράτη-μέλη και οι επιτιθέμενοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και κοστίζουν πάρα πολύ η έκθεση προτείνει στους ε, εκπροσώπους ε, να εφαρμόσουν το άρθρο 222 της συνθήκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω υποστηρίξει την έκθεση αυτή. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια στο σημερινό διαδικτυωμένο κόσμο. Δεν υπάρχουν όρια στα θέματα αυτά γιατί όχι μόνο οι άνθρωποι και το εμπόριο αλλά και τα κράτη εξαρτώνται από την κυβερνοασφάλεια. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χρήση των ψηφιακών δικτύων είναι ασφαλής και ότι οι υποδομές είναι σύμμορφες με τις ανάγκες προστασίας του, των υποδομών αυτών. Θα πρέπει να έχουμε κοινού τρόπους δράσης λοιπόν και να προστατεύσουμε τα δίκτυά μας και θα πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια σε μια τέτοια προστασία και πρέπει να σκεφτούμε και τους νέους και τους εφήβους που χρειάζονται και αυτή η προστασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέπο. Η κυρία Μακοβέ, <clears throat> Τον Μάρτιο 2011 το Κοινοβούλιο υπέστη μια επίθεση στον κυβερνοχώρο. Πριν από μια εβδομάδα η Επιτροπή ήταν και αυτή θύμα παρόμοιες επίθεσης. Επειδή στον κυβερνοχώρο και κατά των διοικήσεων, των κυβερνήσεων, των ε, στρατιωτικών ε, οργανώσεων κλπ. γίνονται αντικείμενο παρόμοιων επιθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προετοιμάσουμε τις υποδομές μας με κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ε, επιθέσεις ε, και επίσης χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία σε ε, δικαστικό επίπεδο για να μπορέσουν να διωχθούν οι δράστες. Υπάρχει ανάγκη από μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παράλληλα με την ασφάλεια και άμυνα, το συστήμα ασφάλειας και άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης να πω ότι το κυβερνοέγκλημα ε, αφορά και τους ε, ιδιώτες χρήστες ε, των συστημάτων αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Μορκουνάιτη Μικουλένινιε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, είχαμε πολλές ε, περιπτώσεις, στις οποίες ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών υπέστησαν επιθέσεις. Η Εστονία, παραδείγματο χάρη, το 2007, όλοι αντιλαμβάνονται πως ο αριθμός αυτών των επιθέσεων θα αυξηθεί, οπότε τα μέτρα τα οποία προτείνει το Κοινοβούλιο είναι επίκαιρα και αναγκαία. Πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράση σε κάθε χώρα έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε στην ε, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας. Κάποιες χώρες οι οποίες δεν είναι και πολύ δημοκρατικές προσπαθούν ε, να χρησιμοποιήσουν με τρόπο λανθασμένο τους υπολογιστές. Δεν πρέπει να ε, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και να χρησιμοποιούνται για πολιτικό σκοπό. Σας ευχαριστώ κυρία Μαρκουνάιτε Μικολίνγε. Ακολουθεί ο κύριος Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ υπερψήφισα την ε, έκθεση αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συγκήτρια για το πάρα πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Ε, πρόκειται βέβαια για πράγματα τα οποία δεν ξέραμε καν στο παρελθόν. Τώρα όλοι μιλάνε για κυβερνοεπιθέσεις, κυβερνοασφάλεια, κυβερνοτραμπουκισμό. Και πρέπει να το δούμε αυτό επίγοντος γιατί όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και απειλούν τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Η δυσκολία λοιπόν είναι το πώς θα ε, το ρυθμίσει αυτό το κράτος ε, όσον αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, πώς θα ρυθμίσει τον ιδιωτικό τομέα και πώς θα ορίσει προδιαγραφές ασφαλείας και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση διότι τα βασικές απειλές ε, προς τα κράτη-μέλη δεν είναι ε, κλασικού χαρακτήρα. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν μια πολύ σημαντική απειλή και οδηγούν σε αποσταθεροποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει μια πολιτική ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο για την πρόληψη παρόμοιων δράσεων. Πρέπει να δημιουργήσει ε, μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από τους ε, καλύτερους εμπειρογνώμονες ε, των κρατών μελών, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τους εμπειρογνώμονες των του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Ρουμανία έχει ξεκινήσει μια τέτοια εργασία προκειμένου να καταπολεμηθεί ε, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και οι επιθέσεις σε αυτόν. Έχουμε λοιπόν ανθρώπινους πόρους, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Κλείσουμε με την έκθεση κλίμα και έρχομαστε στην έκθεση Τάραντ με την κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση, αν και υπάρχουν διάφορα στοιχεία που μπορούν να βγουν αμφιβολίες τώρα. το θέμα της ε, ενεργειακής ασφάλειας ε, γίνεται ένα στοιχείο της ε, πολιτικής ασφάλειας. Να ετονίσω επίση δύο θέματα τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας ε, συχνά εμφανίζεται όταν ε, γίνονται κάποιες ε, φυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τόσο η πολιτική πτυχή όσο και η στρατιωτική. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση περιέχει, λαμβάνει πολλά σημαντικά και σκόπιμα στοιχεία. Επίσης να αναφέρω τον κώδικα καλής συμπεριφοράς που υπάρχει την προστασία του περιβάλλοντος και την επιρροή στην ασφάλεια. Πρόκειται για το σχέδιο Go Green που τονίζει το θέμα της ανεργικής ασφάλειας και πλησμενικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νικολά. Κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στον κόσμο. Ο κύριος Τάραντ αξίζει τους επένους μας για την πολύ σημαντική του εργασία που έχει δείξει τις απόρριες που μπορούν να προκύψουν από τη κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και η οικονομική κρίση. Θα υπάρξουν επιπτώσεις σε επίπεδο ένδυας σε κόσμο, ιδίως στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτές τις επιπτώσεις. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που απειλούνται περισσότερο να την ευκαιρία να προετοιμαστούν καλύτερα και να προστατευτούν και οι πιο ασθενείς είναι οι γυναίκες και τα παιδιά που χρειάζονται την προσοχή μας. το μήνυμα αυτής της έκθεσης σε σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να λάβει αυτό το θέμα στα σοβαρά. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέπο. Ακολουθεί η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Κλιματική αλλαγή και φυσικές ε, καταστροφές έχουν επιπτώσεις στην ειρήνη και την σταθερότητα. Έχουν επιπτώσεις στην οικονομία αλλά είναι και πηγές αστάθειας το, η έλλειψη ύδατος μπορεί να οδηγήσει σε μεταναστευτικά κύματα. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, όλα αυτά τα στοιχεία που και στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της αλλά και στα διάφορα εργαλεία της. Ρεζόμαστε κάποιον ε, εκπρόσωπο για θέματα ε, κλιματικής ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω γραφειοκρατία. Νομίζω ότι η ασφάλεια του κλίματος θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί με στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Υπερψήφισα την ε, έκθεση διότι μέχρι τώρα οι κλιματικές αλλαγές και οι συνέπειές τους εξετάστηκαν μόνο από οικονομικής πλευράς και περιβαλλοντικής αλλά αποτελούν και ένα πρόβλημα για την ασφάλειά μας. Οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν εφαρμόζουμε κάποιες πολιτικές σε εθνικά επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω μελέτες να γίνουν αναφορικά με τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και των ε, φυσικών καταστροφών. Θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφών στο διάλογο με τους βασικούς μας εταίρους. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για περιπτώσεις ε, φυσικών καταστροφών και αυτό μόνο με μέσω μιας βιώσιμης ε, ε, περιβαλλοντικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με την έκθεση Τάραντ. Περνάμε στην έκθεση για Κονσάρι. Θα πω ο κύριος Μέρφυ για δύο λεπτά γιατί μιλάει για εξ ομάδας του. Ευχαριστώ. Όσοι θεωρούν ή λένε πω η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν βελτιώνεται, πρέπει να σημειώσουν τη δήλωση πριν από δύο ημέρε του επισήμου προσώπου του Γενικού Εισαγγελέα, όπου κατηγορείται η μη εγγεγραμμένη αντιπολίτευση ως ε, εξτρεμιστές και κατά για να απαγορευτεί, να απαγορευτούν τα κόμματα, όπως επίσης και οι εφημερίδες Ρεσπούμπλικα και Βίσκλετ ο δορυφορικός σταθμός και η Πλάση και πάρα πολλά site στο ίντερνετ. Είναι σαφές πως η κατάσταση στο Καζακστάν ε, πάει από το κακό στο χειρότερο. Με την απαγόρευση ουσιαστικά ε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ το Καζακστάν θα περάσει άλλον ένα γύρο συλλήψεων και φυλακίσεων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Επιπλέον, ο Βλαντιμίρ Κοσλόφ, επικεφαλή του κόμματος αντιπολίτευση ΑΛΓΑ, ε, ο οποίο καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλάξη, έχασε την έφεσή του πριν από τρει μέρε Το Human Rights Watch είχε πει πω ε, η καταδίκη του βασίζεται σε γενικόλογες κατηγορίε και δεν συμφωνεί με συμβάσει που έχει υπογράψει το Καζακστάν. Επιπλέον, ένα γνωστό αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζει φυλάξη 14 ετών. Απευθύνω έκκληση σήμερα για την άμεση διακοπή των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Συνεργασίας αν δεν βελτιωθούν άμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και αμνηστία άνευ όρων των πολιτικών κρατουμένων. Ζητώ από το διεθνέ Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κοινωνία των Πολιτών να συνταχθούν με αυτή την έκκληση και από την Κάθριν Άστον, η οποία θα πάει στο Καζακστάν την ερχόμενη εβδομάδα, να ξεχαρίσει πως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το καθεστώς Ναζαρμπάγεφ. Είναι απαράδεκτο τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενεργειακούς πόρους του Καζακστάν να προηγούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Μέρφυ. Η κυρία Νικολάη δεν την βλέπω πλέον. Ο κύριος Μπίαλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καζακστάν είναι μια ευκαιρία για αμοιβαία ωφέλη, ιδίω αν λάβουμε υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το Καζακστάν στον παγκόσμιο ενεργειακό χώρο. Θα πρέπει να θυμόμαστε είναι όμω κάτω από την ε, οικονομική επιρροή τη Ρωσία στο Καζακστάν. Επομένω, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε τη χώρα αυτή κοντύτερα στην Ευρώπη. Μια συνεργασία και μια ε, σχέση εταιρικού χαρακτήρα θα φέρει το Καζακστάν κοντύτερα στην ευρωπαϊκή οικονομική σφαίρα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όμω επίση το Καζακστάν να μπει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το ταχύτερο δυνατόν. Η εμπορική αυτή η συνεργασία θα πρέπει να λάβει υπόψη και πράγματα όπω η καλή, δημοκρα... καλή διακυβέρνηση, η δημοκρατία και το κράτο του δικαίου, γιατί αυτέ είναι αρχέ τι οποίε υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Καζακστάν είναι πολύ σημαντικό επίση να διευκρινίσει την κατάσταση τη Κασπία. Αυτό έχει επιπτώσει τη συνεργασία του με άλλε χώρε στην Κεντρική Ασία και πρέπει να βρούμε μια λύση για όλα αυτά τα θέματα των ταχύτερων δυνατών. Πώς στηρίζει το ψήφισμα λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μπιέλεν. Ακολουθεί ο κύριος Κούκαν. Δεν τον βλέπω όμως. Οπότε ακολουθεί η κυρία Μακοβέη την οποία βλέπω. Το 2011 το Καζακστάν έφτασε μόνο σε επίπεδο 2,11 στο δίκτυ αντίληψης διαφάνειας η οργάνωση Freedom House αναφέρει ότι το Καζακστάν εξαρτάται για το δικαστικό σύστημα απόλυτα από την εκτελεστική εξουσία και υπάρχει διαφθορά. Οι δίκες για τα γεγονότα στο Χόζεν περιλαμβάνανε χρήση βίας, εκφοβισμού, βασανιστήριων και χαλκευμένες κατηγορίες η σχέση μας με το Καζακστάν πρέπει να βασίζεται στην πρόοδο στην πολιτική μεταρρύθμιση. Το να αντιμετωπιστεί η διαφθορά στο δικαστικό τομέα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Ο έλεγχος επίσης των σοφρονιστικών ιδρυμάτων θα πρέπει να ξαναγυρίσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και οι πολιτικοί κρατούμενοι θα πρέπει να απελευθερωθούν. Χρειαζόμαστε ε, δεσμευτική ε, αποδοχή αυτών των όρων από το Καζακστάν θα πρέπει να είναι έτοιμο να προχωρήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με σαφείς μηχανισμούς ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Ο κύριος Στάνοκ τώρα. Το Καζακστάν είναι μεγαλύτερο από τη Δυτική Ευρώπη και εκπροσωπεί μια νευραλική χώρα της Κεντρικής Ασίας και είναι μια χώρα που υπάρχει σεβασμός και ανεξιθρησκεία ο ορυκτό πλούτο του Καζακστάν και το μέγεθό του είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αγνοήσει. Είναι μια γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ασία. Σίγουρα πρέπει να αφήσουμε το Καζακστάν να είναι τμήμα, να έχει σχέση με τη Ρωσία ω τμήμα τη ευρωασιατική συνεργασία, αλλά θα πρέπει να έχει στερότερου δεσμού με την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι θα υπάρξουν απτά ωφέλη και για τι δύο πλευρέ που θα πρέπει να συμβαδίζουν με περισσότερη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα για τον λαό του Καζακστάν. Πρέπει να βοηθήσουμε επίση την κυβέρνηση του Καζακστάν να αναπτύξει τις υποδομές της. Αν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η συμφωνία εταιρική σχέση και η προσέγγιση του Καζακστάν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα οδηγήσουν σε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε πολυμερείς οργανισμούς όπου ανήκει το Καζακστάν. Και θα δώσει και μεγαλύτερη ευμάρεια στο λαό της. Γι' αυτό υποστηρίζω την εκθέση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το Καζακστάν είναι μία από τις πλέον σημαντικές χώρες στην περιοχή. Έχει πολύ σημαντικούς ε, πόρους, ε, φυσικούς πόρους ε, και Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μα. Θα ήθελα να παρατηρήσω την σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα αυτή τα τελευταία 20 ετία. Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πρόοδο. Ε, χρειάζεται όμως να δώσουμε και έμφαση και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο μπορούμε να το πράξουμε, διότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν το κάνουν. Το Καζακστάν έχει πολλές ε, συμφωνίες οικονομικές και εμπορικές με την ε, Ρωσία. Θα ήταν καλύτερο να προσελκύσουμε το Καζακστάν περισσότερο μέσω των πολιτικών μας. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με την έκθεση για κονσάρι. Περνάμε τώρα στην έκθεση Φερέρα. Η κυρία Μακοβέη δεν είναι εδώ. Ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, τελευταία φορά με ακούσετε σήμερα και πάλι χαίρομαι που μπορώ να στηρίξω αυτές τις προτάσεις. Βλέπω πως υπήρχαν 474 βουλευτές που υπερψήφισαν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και ικανοποιητικό. Και βεβαίω ε, είναι σημαντική αυτή η έκθεση τη αφορά και την αλληλεία μικρή κλίμακα και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη προστασία. Ειδικά ε, στο μέλλον ε, όσον αφορά την διακρισή που υφίστανται από τα μεγάλα πλοία εργοστάσια που δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους αλλιεύματα και κάνουν και άλλες αθέμητες πρακτικές. Έχουμε άρα διάκριση βάρος των μικρότερων αλλιέων. Προφανώς μειώνονται τα αποθέματα και θα πρέπει να α, τους δώσουμε καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Τελειώσαμε την έκθεση Φερέιρα. Περνάμε στην έκθεση Λέβιν. Κυρία Μακοβέη έφυγε. Να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα γιατί υπάρχει εξωτερική διάσταση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Είναι πολύ περίπλοκη πολιτική και πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προωθήσουμε την αηφορία της αλληλείας και της βιοπικιλότητας, αλλά βεβαίως μπορούμε να βελτιώσουμε την διαχείριση της διεθνούς αλίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντονίσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εναρμονισμένη πολιτική και να ακολουθήσουμε συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες. Επίσης θα πρέπει να δούμε το σημαντικό ρόλο που παίζει η Ένωση στην καταπολέμηση της ε, λαθραλίας και παράνομης αλίας. Είναι σημαντικό αυτό για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου και περνούμε τώρα στην τελευταία έκθεση για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014. Η κυρία Μακοβέη δυστυχώς δεν είναι παρούσα, αλλά η κυρία Μπασέσκου ευτυχώς είναι παρούσα. Έχω ψηφίσει υπέρ του ψηφίσματος, λέει η κυρία Μπασέσκου γιατί πιστεύω ότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν επίσης θα πρέπει να βασίζεται η σύνθεσή της και σε δημοκρατικές αρχές και αυτό σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την εκλογή του να εκφράσει την άποψή του για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποστηρίζεται από πολιτικά κόμματα. Χρειάζεται όμως να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες και να, στην Κομισιόν και να δίνουμε τη δυνατότητα να προταχθούν οι εκλογές για ένα μήνα. Με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν θα μπορέσει να αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερο έλεγχο για την Κομισιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και κλείνουμε με την κυρία Σίνκλα. Κύριε Πρόεδρε, σε καιρούς λιτότητος οι πολίτε μου δεν θέλουν να σπαταλούνται τα χρήματά του για πολιτική προπαγάνδα και εκστρατείε. Εγώ καταψήφισα όλε αυτέ τι προτάσει, οι οποίε θέλουν να υποστηρίξουν τα πανευρωπαϊκά κόμματα για να διαδώσουν την ιδεολογία του φεδεραλισμού σε όλη την Ευρώπη. Οι περισσότεροι πολίτε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρούν ότι έχουν μια ταυτότητα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Έχουν εκφράσει την απόρριψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκλογέ και οι δημοσκοπήσει το έχουν καταδείξει αυτό και έχουν τονίσει οι πολίτες μου ότι θέλουν ένα δημοψήφισμα. Δεν θέλουν άλλη προπαγάνδα που να πληρώνεται από του φόρου του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε περικοπέ σε δημόσιες υπηρεσίες όσο δίνουμε όλο και περισσότερα λεφτά στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Θέλουμε το 2014 να υπάρξει ένα δημοψήφισμα και αυτό θα επιτρέψει στους εκλογείς του Ηνωμένου Βασίλειου να στείλουν το σωστό μήνυμα στην κυβέρνησή μας ότι θέλουμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε μέσα ή έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κυρία Σίνκλερ. Κλείσαμε και με τις επεξηγήσεις ψήφου στο τελευταίο θέμα της εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κλείνουμε λοιπόν και την ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασής μας. Συνεχίζουμε πάλι στις 3 και σας εύχομαι καλή όρεξη.